Συνόδου. Ο κύριος Λαουρέντσιου Ρεμπέκα από, ε, ε εγκατέλειψε την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και προσεχώρησε στην ομάδα ΙΕΝΕΦ. Ο κύριος Χουάν Φερνάντο Λόπες Αγγουιλάρ στις 22 Ιουλίου 2015 προσεχώρησε στην